Από ό,τι βλέπω, όχι επομένω ε, εγκρίνονται. Λοιπόν, Οι Ισπανικέ Αρχέ με ενημέρωσαν ότι η κυρία Άλβαρε πρόκειται να αντικατασταθεί τον κύριο Σέρχιο Κουτιέρε Πριέτο. Αυτό θα λάβει την βουλευτική έδρα με ισχύ τη πράξη αυτή από τι 19 Ιουλίου του 2010. Καλώ όρισε ο νέο συνάδελφο. Δεν ξέρω αν παρίσταται. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν παρίσταται. Θα έχασε το δρόμο. Θα μάθει, θα μάθει. Τώρα, δυνάμει του άρθρου 2, παράγραφος 2, ε, θα πρέπει να κάνουμε την εξακρίβωση της εντολής. Και θα πρέπει να περιμένουμε μήπως υποβληθεί κάποια τυχόν ένσταση κατά ε, της κατάληψης έδρας από τον κύριο Κουτιέρης Πριέτο. Οπότε με αυτή την επιφύλαξη θα αποτελέσει τακτικό μέλος του Κοινοβουλίου, όμως πρόκειται να υποβάλει κάποια δήλωση ότι δεν έχει αναλάβει κάποια άλλα καθήκοντα, κάποιο άλλο λειτουργήμα που να αντιβαίνουν με το λειτουργήμα του Ευρωπαίου Βουλευτού. Επίσης, έχουμε την κυρία Ανιές Άγκης, η οποία αποτελεί το αντικείμενο αίτησης άρσης της ε, βουλευτικής ασυλίας διότι έχει εμπλακεί σε κάποια δίκη ε, εναντίον της στην Βουδαπέστη.